Κυρίες και κύριοι, πριν από ένα έτος ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη, η οποία έφερε ελευθερία σε πολλούς από τους νότιους γειτονές μας και στη Συρία. Οι άνθρωποι έχουν βγει στους ε, δρόμους, διαδήλωσαν ειρηνικά, γεμάτη ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Ε, και αυτό το οποίο ζούμε είναι πως ένας κτηνόδης δικτάτορας αποφάσισε να διεξάγει ανοιχτό πόλεμο εναντίον του λαού του και κατά της ίδιας ελευθερίας. Πάνω από 8.000 άτομα έχουν πεθάνει ήδη φέτος στην Συρία και η ματοχυσία δεν τελειώνει. Οι άνθρωποι στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο, όλοι μας, είμαστε αν και άναβη μπροστά στην απάνθρωπη κτηνοδία του καθεστώτος, και του καθεστώτος αυτού και την αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να το σταματήσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση στον πρόεδρο Αλ Ασάντ τουλάχιστον να επιτρέψει πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια για τον άμαχο πληθυσμό. Και οπωσδήποτε θα συμφωνείτε μαζί μου στην έκκλησή μου προς τη διεθνή κοινότητα, τον ΟΗΕ, την, ε, τον Αραβικό Σύνδεσμο και τον πρόσωπό του στον ε, Κόφι Ενάν για να υπάρξει μια ειρήνη στην περιοχή. Επίσης απευθύνουμε έκκληση στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχουν ε, δικαίωμα βέτο να μην εξαρτούν την στάση τους από διάφορα συμφέροντα. Χτες, κυρίες και κύριοι, είχαμε για πολλωστή φορά την 11η Μαρτίου. Όπως ξέρετε, 11 Μαρτίου 2004 είχαμε στη Μαντρίτη ε, το τρομακτικό τρομοκρατικό χτύπημα ε, σε ευρωπαϊκό έδαφος με 119 νεκρούς και 1.800 τραυματίες. Τιμούμε όλα τα τμήματα της τρομοκρατίας από, το Μαδρίτη, από τη Μαδρίτη μέχρι το Λονδίνο και την Μπολόνια. Εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στεκόμαστε στο πλάι των οικογενειών που επλήγησαν από αυτές τις φρικτές πράξεις. Στεκόμαστε στο πλάι όσων έξαν συγγενείς και φίλους και αυτές τις στιγμές σκεφτόμαστε και τους επιζώντες τρομοκρατικών επιθέσεων όμως για το υπόλοιπο της ζωής τους θα υποφέρουν από τα ψυχολογικά και σωματικά τραύματα που τους άφησαν αυτές. Και βεβαίω απορρίπτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε μορφή τρομοκρατίας με τη δειλή ανωνυμία της. Η τρομοκρατία αποτελεί μία από τις πιο αποκρουστικές μορφές βίας της σύγχρονης εποχής. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους επιζώντες και τα θύματα της τρομοκρατίας. Χτες και η Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, όπως και όλοι εμείς, τίμησε την επέτειο της ε, καταστροφής του τσουνάμι του 2011. Θυμόμαστε όλοι τις εικόνες αυτής της τρομερής τραγωδίας και της πυρηνικής καταστροφής που ακολούθησε το τσουνάμι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης το πρώτο σημείο του σήμερα θα ασχοληθεί με το γεγονός αυτό και τις συνέπειες του όμως ήδη στην αρχή της σημερινής μας συνεδρίασης θα ήθελα να εκφράσω την συμπόνια μας για τα πάρα πολλά θύματα αυτής της φυσικής καταστροφής και της πυρηνικής καταστροφής. Θα ήθελα επίσης να σας παρακαλέσω να σηκωθείτε και για τα θύματα στην Συρία και τα θύματα της τρομοκρατίας και αυτής της φυσικής καταστροφής για ένα λεπτό σιγής.